So we start. Point one Αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα. Ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Το πρώτο σημείο είναι η έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Ήθελα να σας ενημερώσω σε σχέση με την ημερήσια διάταξη ότι το σημείο 7, ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με την Καμπότζη, θα γίνει κυκλισμένο των θυρών. Δεν έχω λάβει κάποια άλλη έτοιμα σε σχέση με την ημερήσια διάταξη. Αν δεν έχετε αντίρρηση να θεωρήσω ότι εγκρίθηκε. Σημείο 2, όπως συνήθως, να ανακοινώσεις του Προέδρου μεταδίδεται μέσω ίντερνετ τη συνεδρίαση. Καλημερίζω όλους από τη Λισαβόνα μέχρι το, το, το Τάλιν και τη Θεσσαλονίκη. Επίσης υπάρχει, προσφέρεται διερμηνία στη συνεδρίαση αυτή και διερμηνεί σα παρακαλούμε να μιλάτε καθαρά και σχετικά αργά. Θα ήθελα να καλωσορίσω πίσω στην κυρία Στεφανία Ναρτέλη στη γραμματεία της Επιτροπής μας. Ξεκίνησε αυτό το μήνα. Καλώς ήρθατε. Σημείο 3 διαπραγματεύσεις σε εξέλιξη. Μία έχουμε αυτή τη στιγμή. Είναι screening για άμεσες ε, ξένες επενδύσεις. Εισηγητής ο κύριος Προύστ. Τη θέση της Επιτροπή είναι τα την ε, υπερψήφισε το Μάιο. Προχωρούν οι διαπραγματεύσεις κάπως αργά, βρισκόμαστε σε πρώτες φάσεις, στις αρχικές φάσεις, ζητούμε ζητήματα διαδικαστικά. Η πρώτη συνάντηση έγινε στις 27 Σεπτεμβρίου και η δεύτερη αύριο, 11 Οκτωβρίου. Βεβαίω αυτά που θα συζητηθούν κατά προτεραιότητα είναι αυτά που, τα θέματα για τα οποία υπάρχουν πολιτικές διαφορές, διαφορές. Θα προσπαθήσουν και ο συντονιστής και οι υπόλοιποι να βρεθεί μια συμβιβαστική λίστη πριν τα Χριστούγεννα. Και να γίνει και, άλλη, και άλλες συναντήσεις διαλόγου και με το Συμβουλίο τέλη Νοεμβρίου. Έχετε κάποια παρατήρηση, όχι. Θα συνεχίσω λοιπόν με τα σημεία 4 και 5. Θα τα εξετάσουμε από κοινού για τις ε, συμφωνίες εμπορίου με την Ιαπωνία. Βρισκόμαστε στη διαδικασία επικύρωσης. Πρέπει να δώσει τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο. Η προθεσμία για τροπολογίας ήταν η 2 Οκτωβρίου. Όπως ήθιστε θα δώσω το λόγο στον ε, εισηγητή μας, τον κύριο Περέιρα. Δεν είναι εδώ όμως, ο κύριος Μάρτιν θα το αντικαταστήσει, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καλημέρα. Πριν μιλήσω εκ μέρους του Πέντρο, θα ήθελα να μιλήσω ε, εξ ονόματός μου και να συγχαρώ τον Πέδρο για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τη συζήτηση και συνέχισε μέχρι το τέλος της διαδικασίας να πιέζει την πλευρά της Ιαπωνίας για ζητήματα που θεωρεί σημαντικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα μιλώ εξ του Πέδρου. Ζητά συγγνώμη που δεν μπορώ να παρευρεθώ για να συζητήσουμε την εξέταση των τροπολογιών που έχουν υποβληθεί επί της εκθεσής μου για την, ε, οικονομική, για, την εμπορική συμφωνία με την Ιαπωνία, αλλά ε, πρέπει να συμμετάσχω σε μια αντιπροσωπεία οικονομικής συνεργασίας με την ε, Ιαπωνία. Ο πρέσβης μας έστειλε επιστολή με τις οποία μας ενημερώνει ότι η πρώτη συνεδρίαση θα γίνει τον Οκτώβριο των Αρμοδίων Υπουργείων εκτιμούμε αυτό το βήμα. Θεωρώ ότι η συμφωνία αυτή είναι σημαντική για τρεις λόγους. Πρώτον, η εμπορική συμφωνία με την Ιαπωνία έχει μεγάλη στρατηγική ε, σημασία, ε, ιδίω αυτή τη συγκυρία, γιατί δείχνει ότι υποστηρίζουμε το ελεύθερο εμπόριο με βάση τους διεθνείς κανόνες και αντιτιθέμεθα στην προστατευτική ε, προσέγγιση του Τραμπ. Δεύτερον, γιατί έχει μεγάλη, ε, ε, επίσης έχει μεγάλη σημασία στην περιοχή. Δεύτερον, θεωρούμε ότι είναι ισορροπημένη από οικονομικής απόψεως, δίνει τη δυνατότητα σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση στην ιαπωνική αγορά και ταυτόχρονα προστατεύει τους ευαίσθητους τομείς. Και τρίτον, και πλέον σημαντικό, είναι μία από τις συμφωνίες νέας γενιάς, από αυτές που συμπεριλαμβάνουν ρήτρε για την προστασία του περιβάλλοντος και των εργατικών δικαιωμάτων. Είναι η πρώτη τέτοια συμφωνία που ε, σύμφωνα και με τη διακήρυξη των Παρισίων υπάρχει μια, υπάρχει μια αναφορά μάλλον στη διακήρυξη των Παρισίων και επίσης στην ε, εταιρική κοινωνική ευθύνη και ένας μηχανισμός παρακολούθησης των διατάξεων αυτών. Θα ήθελα να ευχαριστώ, στήσω τους συναδέλφους για την συνεισφορά τους. Έλαβα 2003, ε, συγγνώμη, 236 τροπολογίες με τους συναδέλφους από τους σοσιαλιστές υποβάλαμε 18. Οι περισσότερες από αυτές έχουν σχέση με τη διόρθωση στοιχείων για παράδειγμα ο αριθμός των πόλεων που θα ε, ε, εμπλακούν σε διαδικασίες δημοσίες ε, προκηρύξεων. Στην τροπολογία 134, για παράδειγμα, αναφερόμαστε στην απόφαση της Ιαπωνίας να δημιουργήσει μια επιτροπή διυπουργική για την βιώσιμη ανάπτυξη και αυτό έγινε μετά τη σύνταξη της έκθεσης. Εκτός αυτού υπάρχουν και τροπολογίες με τις οποίες προσπαθούμε να εισάγουμε θέματα σημαντικά που δεν μπορούσαμε αρχικά να βάλουμε για λόγους χώρου. 103 για τα ζητήματα του φύλου, 218 για τη συνεργασία που θα πρέπει να υπάρξει με την Ιαπωνία σε παγκόσμιο επίπεδο για την προώθηση του ελευθέρου εμπορίου στο πλαίσιο των συμφωνιών του ΠΟΕ και επίσης το 2027 για την παρακολούθηση των, ε, εσωτερικών θεμάτων. Μετά θα μπορούσα να ομαδοποιήσω τις τροπολογίες ως εξή. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν εκείνες οι οποίες προσθέτουν στοιχεία και με τις οποίες σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι συμφωνούμε. Δεύτερον, είναι οι τροπολογίες της παραγράφου 11 που αναφέρονται περισσότερο στο ευαίσθητο θέμα της ρήτρα της βιώσιμης ανάπτυξης. Και τρίτον, η ομάδα εκείνη των τροπολογιών με τις οποίες δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα μπορούσαμε να τις δεχτούμε. Καταλήξαμε σε 22 συμβιβαστικές τροπολογίες και θα τις παρουσιάσω στους σκιώδες, τις παρουσίασα μάλλον στους σκιώδες και προσπαθήσαμε να έχουμε στις 8 Οκτωβρίου το απόγευμα μια επικοδομητική συζήτηση Συζητήσαμε τις συμβιβαστικέ και προσπαθήσαμε κυρίως να βρούμε μια συμβιβαστική λύση για την παράγραφο 11 που όπως σας είπα είναι εκείνη που αναφέρεται στη βιώσιμη ανάπτυξη. Θα έλεγα ότι αυτή η πρώτη συνάντηση των σκιωδών πήγε καλά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους. Και κλείνει ο κύριος Περέιρα λέγοντας ότι προσβλέπω στη συνεργασία μας και να σας ξαναδώ όλους στην επόμενη συνάντηση των σκιωδών. Σε ευχαριστώ, Ντέιβι. Θα δώσω τώρα το λόγο στους κοιόδης εισηγητέ για τρία λεπτά στον καθένα από το ΕΛΚ. Ο κύριος Χάνσεν είναι ο πρώτος. Ναι, ευχαριστώ και καλημέρα. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον συνάλφο Σίλβα Περέιρα για την πολύ καλή του μέχρι τώρα δουλειά. Εξεργαζόμαστε τώρα συμβιβαστικές προτάσεις επί των τρόπολογιών που μόλις παρουσίασε ο κύριος ε, Μάρτιν. Θέλω επίση να ευχαριστήσω και τον κύριο Βαλένσα, με τον οποίο συγκαταθέτω αρκετέ τροπολογίε. Ήταν ο σκιώδη συγητή, τώρα είμαι εγώ στη θέση του. Υπάρχουν διάφορα σημεία που εκκρεμούν ακόμη. Ο κύριος Μάρτιν ανέφερε ένα από τα σημαντικότερα, τα σημεία 10 και 11, όπου αναφέρονται κυρώσεις. Θέλουμε να είναι αποτελεσματικό το σύστημα, αλλά για την επιβολή των κυρώσεων ε, δεν έχουμε καταλήξει. Είχαμε τη Δευτέρα την πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Η Ιαπωνία νομίζω ότι έχει δείξει ότι δεσμεύεται και ε, θέλει να υλοποιήσει σωστά τη συμφωνία. Μιλήσατε και για την επιστολή του πρέσβη Κουντάμα. Και αυτό είναι ένα σαφές μήνυμα κατά την απόψή μου και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχει μεταρρυθμίσει την εργατική νομοθεσία ε, για πρώτη φορά μέσα σε 70 χρόνια η Ιαπωνία, άρα υπάρχουν συγκεκριμένα βήματα από πλευράς της χώρας και θα συνεργαστούμε μαζί με τον εισηγητή για το θέμα αυτό. Δι, έχουμε, πιστεύω, πετύχει αρκετά. Ο στόχος είναι να έχουμε περατώσει μέχρι τα τέλη της θητείας ε, το ζήτημα και αισιοδοξία υπάρχει αν δει κανεί την πρόοδο που έχουμε ήδη επιτύχει. Ο κ. Καμάλα από το ECR. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον εισηγητή και τους κοιόδης εισηγητές. Τον εισηγητή θέλω να τον ευχαριστήσω για την ισορροπημένη του έκθεση πρώτα απ' όλα, που αναφέρει πολλά από τα επιτεύγματα αυτής της συμφωνίας. Πολλές φορές οι εκτιμήσεις πέφτουν έξω ε, και εγώ είχα ε, κάνει λάθος εκτιμήσεις, δεν περίμενα τόσες πολλές τροπολογίες. Ε, φαίνεται όμως ότι υπάρχουν ανησυχίες από πολλούς και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Υπάρχουν πάντως θετικές συνεισφορές που δείχνουν ε, ότι υπάρχουν, υπάρχει ωφέλη και για τις δύο πλευρές ό,τι αφορά τον όγκο των συναλλαγών και νομίζω ότι υπάρχουν και άλλες τροπολογίες που μιλούν για την κατάργηση δασμών στα ε, περισσότερα αγαθά, την άρση των μη δασμολογικών δασμών, άνοιγμα της αγοράς δημοσιοπρομηθειών της ε, Ιαπωνίας, η παροχή υπηρεσιών, μη διακρίσεις κτλ. κτλ. Σίγουρα ε, οι υπηρεσίες έχουν ε, μεγάλη σημασία ε, και στον τομέα της γεωργίας και της μεταποίησης. Εμείς θεωρούμε ότι αυτή η οικονομική συμφωνία θα στηρίξει και το δίκαιο ελεύθερο εμπόριο και η βιώσιμη διάσταση έχει προσλάβει σημασία. Έχουμε το κεφάλαιο εμπόριο, βιώσιμη ανάπτυξη και νομίζω ότι και οι δύο πλευρέ εκφράζουν τη δέσμευσή του στη Συμφωνία των Παρισιών. Χαίρομαστε επίση που κάποιε τροπολογίε μιλάνε για την εταιρική διακυβέρνηση, τα ΕΣΜΜΕ και τα ωφέλη από τη Συμφωνία για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, που ξέρουμε ότι αντιπροσωπεύουν πολύ μεγάλο μερίδιο εταιριών που εξάγουν προς την Ιαπωνία. Ελπίζουμε αυτό να μην ε, θεωρηθεί ως μια ε, επιχείρηση για τις μεγάλες μόνο επιχειρήσεις, αλλά μια συμφωνία που θα ωφελήσει όλες τις επιχειρήσεις. Επίσης αντιλαμβανόμαστε το ζωτικό ρόλο των διασυνοριακών ροών δεδομένων. Όσοι εργάζονται στο μέσο τεχνολογίας και άλλους κλάδους αναγνωρίζουν ότι τα δεδομένα είναι το νόμισμα των ημερών. Σε ό,τι αφορά τώρα τη βιώσιμη ανάπτυξη, το σχετικό κεφάλαιο. Αυτός ο μηχανισμός ε, για την επιβολή κυρώσεων είναι ένα θέμα που καιρό το συζητάμε και δεν έχει ακόμη υπάρξει συνένεση. Είχαμε στηρίξει κάποιες προτάσεις. Αλλά δεν νομίζω ότι όταν έχουμε απέναντί μας ένα νόμο ιδεατήτερο όπως είναι που έπρεπε να συνεχίσουμε ε, να εφαρμόζουμε το ισχύον σύστημα. Σε ό,τι διαφορά τις διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης και του βιώσιμου εμπορίου. Για να αλλάξουμε, μια, να αλλάξουμε τη στάση και την πολιτική μας, εμείς χαιρετίζουμε σε ένα βαθμό τα όσα λέγονται, αλλά πιστεύουμε ότι αυτά θα πρέπει να βασιστούν στη συνεργασία και το διάλογο. Εν γέννη, μας άρεσε το πρώτο κείμενο. Θα στηρίξουμε αρκετές από τις τροπολογίες και θέλω να ευχαριστήσω τον Σίγητη και τους Σκιώδης. πρόεδρο. σας ευχαριστώ. Να διαχείρισω από την άλλη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. τη περισσότερες από τις τροπολογίες νομίζω ότι δείχνουν ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, ότι είναι θετική δηλαδή αυτή η συμφωνία και θα έχει θετικά αποτελέσματα. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω θερμά τον εισηγητή Σίλβα για την καλή του δουλειά, για την προσήλωσή του στο να προχωρήσει το θέμα και νομίζω ότι είναι επίκαιρο να στείλουμε ένα σοβαρό μήνυμα, θετικό μήνυμα και πρέπει επίσης ε, να γνωρίζουμε όταν σίγουρα υπάρχουν ε, πτυχές ε, που θέλουμε να τις συμπληρώσουμε και είναι θεμητό, υπάρχουν και κάποια βασικά που πρέπει να λυθούν, όμως θέλουμε να είμαστε επικοδομητικοί για να δώσουμε ένα μήνυμα τελικά ότι θέλουμε ένα ελεύθερο δίκαιο εμπόριο και θέλουμε να κρατήσουμε ψηλά εμείς το λάβαρο της Ευρώπης. Ε, η συμφωνία για μένα έχει μεγάλη σημασία. Είμαστε υπέρ ε, ενός εμπορίου που θα βασίζεται σε κανόνες, ε, ε, ελεύθερο εμπόριο, δίκαιο εμπόριο. Και θέλουμε να προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, ό,τι αφορά συγκεκριμένες τροπολογίες, υπάρχουν κάποιες τροπολογίες που είναι αρνητικές. Δεν ξέρω Ξέρουν αυτοί που συνέταξαν τι τροπολογίε αυτέ, ε, οι ομάδε, οι άνθρωποι, οι συγκεκριμένοι βουλευτέ στη χώρα, έχουν πάει στην Ιαπωνία. Ξέρουν ε, ε, τι θα πει σεβασμό προ τον απέναντι, προ τον διαπραγματευτή κτλ. Επίση, θα υπογραφεί μια ευρεία συμφωνία ουσιαστικά σε σχέση με άλλες που είχε υπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά, εμάς μας ενδιαφέρει και η προστασία των ε, προσωπικών δεδομένων, ένα θέμα σημαντικό. Τη ροή δεδομένων θα την παρακολουθήσουμε. Είναι ένα θέμα που μας ενδιαφέρει. Έχουμε και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων και για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό σκηνοβούλιο να παραμένουμε ενήμεροι ε, σε ό,τι αφορά ε, τις ενδεχόμενες αλλαγές. Επίσης, σε ό,τι αφορά το μηχανισμό ISDS, το έχει πει και η Κομισιόν, δεν έχει πλέον εντολή, δεν πρέπει ε, να καταρκωθεί εμπιστοσύνη. Θέλουμε να υπάρχει ένα ελεύθερο εμπόριο ως κοινωνία, ως κοινοβούλιο. Θέλουμε να συνεργαζόμαστε και στη συνέχεια, στη φάση της ε, εφαρμογής, της εκτέλεσης. Και ίσως ε, κάποιες συμβαστικές προτάσεις ε, θα μπορούσαν να δώσουν σημασία και έμφαση στην υλοποίηση, στην εφαρμογή γιατί και θα δούμε ουσιαστικά το πώς ε, θα, ε, ποιος θα είναι ο αντίκτυπος αυτής της ε, συμφωνίας. Πάντως η στάση μας είναι επικοδομητική και θα συνεχίσουμε τη συνεργασία. Ευχαριστώ κύριος Μπούχνερ τώρα εκ μέρους των Πρασίνων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή ο οποίος πραγματικά προσπάθησε να καταλήξει σε ένα συμβιβασμό μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων και χαίρομαι ιδιαίτερω ε, που το αποτέλεσμα είναι τόσο καλό. Σε ό,τι αφορά δε το περιεχόμενο, σε ό,τι αφορά τους Ιάπωνες, σε ό,τι αφορά το χάρι, χάρτη βιώσιμης ανάπτυξης. Δύο παρατηρήσεις. δεν μιλάμε για τους Ιάπωνες μόνο, μιλάμε και για εμάς. Ουσιαστικά πρέπει να έχουμε τα ίδια μέτρα και σταθμά. Πρέπει να έχουμε κάποια πρότυπα. Και ε, θέλουμε να ε, προωθήσουμε το περιβάλλον και την εργατική, εργασιακή νομοθεσία. Το δεύτερο, εγώ είχα εργαστεί ε, στην Ιαπωνία πριν δύο χρόνια και τη γλώσσα την γνωρίζω, άρα δεν ε, δέχομαι κατηγορίες ότι κάποιοι που έχουμε συντάξει τροπολογίες δεν ξέρουμε την χώρα. Σε ό,τι αφορά τις εκπομπές ε, του άνθρακα είναι από τις υψηλότερες στον κόσμο στην Ιαπωνία. 9,5 τόνοι κατά κεφάλι είναι και έχουν αυξηθεί μετά το 1990 το 9% περίπου του συνόλου της ενέργειας στην Ιαπωνία προέρχεται από την καύση, από τα ορυκτά καύση, πετρέλαιο, άνθρακα και όπως είπα, και μεθάνιο βέβαια. Και αυτό δεν χρειάζεται να συμβαίνει. Έχουμε δει μελέτες που λένε ότι θα μπορούσε να μην ισχύει. Και σε ό,τι αφορά ε, την ατομική επίσης ενέργεια ε, υπάρχει πρόβλημα και μπλοκάρεται ε, πάρα πολύ αυτή η ε, πρόοδος. Ε, υπάρχει και το πρόβλημα ε, της υλοτόμησης και αυτό σίγουρα μας ενδιαφέρει και εμάς στην Ευρώπη. Τώρα, θα έπρεπε να υπάρχει ένα κεφάλαιο για το STS και για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Επαναλαμβάνω και για εμάς έχουν ενδιαφέρον όλα αυτά. Τέλος, ό,τι αφορά τους κανόνες, ε, τους οικονομικούς κανόνες, ε, πραγματικά ε, δεν είναι καθόλου καλές, καταστροφικές κατεμές, διότι είδαμε πώς η απελευθέρωση οδήγησε σε κρίση και εδώ βλέπουμε ακόμα περισσότερο τα αποτελέσματα. Ευχαριστώ, Χέλμου του όλους εκ μέρους της ΓΚΟΕ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Φυσικά και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή ο οποίος προσπάθησε να καταλήξει σε συμβιβασμούς. Λόγω του ότι κατατέθηκαν πάρα πολλές ε, τροπολογίες. Άλλες θετικές και άλλες ε, επικριτικές απέναντι στην ε, συμφωνία αυτή. Και προσπαθούμε να βρούμε ένα τρόπο για να ισορροπήσουμε. Αυτό είναι ανοιχτό κατά με αν θα το πετύχουμε. Εμεί σαν ομάδα ήδη εκφράσαμε έντονε επικρίσει ό,τι αφορά την ε, ε, συμφωνία αυτό Ο κύριο Μπούχνερ από του Πρασίνου ανέφερε ορισμένα πράγματα σε ό,τι αφορά τη βιωσιμότητα, το θεματολόγιο της Η εφορία μα ενδιαφέρει. Έχουμε και ε, τους 17 στόχους και τον χρονικό ορίζοντα του 2030 και απότερο ορίζοντας το 2050, σίγουρα αυτοί οι στόχοι πρέπει να επιτευχθούν και εμείς ε, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ενισχυμένος ανταγωνισμός ε, σε ό,τι αφορά τη γεωργική παραγωγή, αλλά και άλλες πτυχές ε, της πραγματικής οικονομίας, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε ακριβώς τι αλληλεπίδραση υπάρχει μεταξύ ανταγωνισμού στην αγορά και δομών παραγωγικών. Δηλαδή δεν μπορούμε να αρνηθούμε ε, ότι ένας κλάδος που έχει πρόσβαση στην αγορά ε, τροφίμων θα απειλήσει ε, την ύπαρξη των μικρών επιχειρήσεων στην Ιαπωνία. Αυτό πρέπει να το δούμε πάρα πολύ προσεκτικά έχοντας υπόψη ναι, και την προσφορά για να μην δημιουργήσουμε δεσπόσες θέσεις. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη και θα πρέπει να είμαστε ειλικρινεί. Μια διμερή συμφωνία δεν μπορεί να αφήνει έξω περιβάλλον, βιομηχανία, κοινωνική δικαιοσύνη, οικονομική ανάπτυξη. Επίσης, αυτοί οι οικονομικοί κανόνες και μας, ε, μας δημιουργούν προβλήματα. σε ό,τι αφορά και την ίδια τη θέση της ε, και την ισχύ της ιαπωνικής οικονομίας ε, υπάρχει, θα υπάρξει μεγάλη πίεση και αυτό το θέμα επίσης της απελευθέρωσης, της φιλελευθεροποίησης. Τρίτον, η παράνομη υλοτόμηση, Επίσης ότι δεν υπάρχει απαγόρευση όταν αναφέρεται ε, το πρόβλημα της φαλαινοθυρίας ε, και του τόνου, του γαλαζόπτερου κτλ. Υπάρχουν διάφοροι τομείς ε, που δεν θα πρέπει να συνεχίσουμε να επιτρέπουμε να συνεχίσουν αυτές τις δραστηριότητες. Επίσης, θέλω να πω ότι όλα αυτά τα θέματα τα οποία αναφέραμε τα συμπεριλαμβάνουμε σε τροπολογίες μας αν δεν περάσουν όλα αυτά θα ζητήσουμε να, να ζητήσει μια δεύτερη επικύρωση αυτής της συμφωνίας. Ευχαριστώ κυρία Μπεγκίνου. Το Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον εισηγητή για την πολύτιμη εργασία του. Όπως έχω πει και στο παρελθόν, εμείς βλέπουμε θετικά αυτή τη συμφωνία που οπωσδήποτε ε, θα βοηθήσει τις ευρωπαϊκές ε, επιχειρήσεις ε, να μπουν σε σημαντικά τμήματα της αγοράς της Ιαπωνίας. Η κατάσταση στη διεθνή αγορά, η χρονική στιγμή είναι πολύ ευαίσθητη και οπωσδήποτε θα πρέπει να βοηθηθούν να προστατευτούν ε, συγκεκριμένοι τομείς όσον αφορά τι δραστηριότητές τους και τις θέσει εργασίας. Θα πρέπει οπωσδήποτε ε, ε, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στην Ιαπωνία να έχουν την ίδια μεταχείριση που έχουν οι ιαπωνικέ στην Ευρώπη. Θα ήθελα να ζητήσω από τον εισηγητή να λάβει υπόψη του και τα στοιχεία τα οποία έχω αναφέρει εγώ όταν, για θέματα όπως είναι ας πούμε η παράνομη διακίνηση Επίση επίσης το γεγονός ότι ε, η Ιαπωνία παρότι είναι προχωρημένη η σύγχρονη χώρα επιμένει και διατηρεί την θανατική ποινή. Ε, επίσης ε, νομίζω ότι πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί έτσι ώστε η προστασία των καταναλωτών σωστά να καλύπτεται και χαίρομαι που αυτή η θέση έχει γίνει δεκτή. Ε, υπάρχει επίσης ε, και μία ε, ρήτρα η οποία προσωμιάζει στη Συμφωνία ΣΕΤΑ και ευελπιστώ ότι η Κομισιόν δεν θα παρουσιάσει μέσα στον επόμενο χρόνο μία συμφωνία αυτού του τύπου. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Για δύο λεπτά τώρα τα μέλη της Επιτροπής. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον ε, Πέτρο, τον εισηγητή μας ε, για, για το προσχέδιο της έκθεσης καθώς επίσης ε, και για τη συνεργασία στα πλαίσια του Monitor Group. θα ήθελα να κάνω κάποια γενικά σχόλια τα οποία καλύπτουν όλες τις τροπολογίες που έχω υποβάλει. Πρώτον, όπως είπε και ο Κλέο Μπίχνερ, σχετικά με την βιώσιμη ανάπτυξη, η τροπολογία μου δεν αφορούν ε, επίκριση προς την Ιαπωνία, αλλά πιο πολύ ε, την ευρωπαϊκή πλευρά των διαπραγματεύσεων, με την έννοια ότι δεν θεωρώ ότι προχωρήσαμε αρκετά Αναφέρθηκε βέβαια ότι υπάρχει διαφορά απόψεων όσον αφορά αρκετά στοιχεία που σχετίζονται με την βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά νομίζω ότι κάθε φορά που έχει ε, ε, παρουσιαστεί το θέμα στην Ολομέλεια, ε, το θέμα έχει περάσει, έχει περάσει μάλιστα και το θέμα που πάει παραπέρα, δηλαδή στις κυρώσεις σε περίπτωση μη εφαρμογής ρητρών για την βιώσιμη ανάπτυξη τρεις φορές ε, μάλιστα ε, στην Ολομέλεια έχουμε περάσει αποφάσεις οι οποίες αφορούν την υποχρεωτική και έναντι κυρώσεων ε, ε, υποχρέωση για, βιώσιμη, για ρήτρες βιώσιμης ανάπτυξης. Επίσης υπάρχει και μία έκθεση για την οποία ήμουν εισηγήτρια για την ε, υλοποίηση της εμπορικής πολιτικής. Εκεί ζητούσαμε να συνεχιστούν οι χειρώσει για, παράνομα, για παράνομες εμπορικές πρακτικές. Ε, όσον αφορά το εμπόριο και την ε, βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι ηρωνικό γιατί εδώ μιλάμε τώρα με την Ιαπωνία που έχουν ε, υπογράψει παρόμοια μέτρα στα πλαίσια του τύπου. Επομένως, εμείς θα πρέπει μαζί με έναν τέτοιον σημαντικό σύμμαχο να προχωρήσουμε έτσι ώστε να καταφέρουμε να, δημιουργού, να συνεχίσουμε στη δημιουργία ε, παγκόσμιας ανάπτυξης και να επανακτήσουμε την εμπιστοσύνη του κόσμου. Ε, δεν υπάρχει ένα σύστημα IDS ε, ή ISS και χαιρόμαστε γιατί σε αυτή την περίπτωση, σε σχέση με την ΣΕΤΑ, θα είναι πιο εύκολη η διαδικασία έγκρισης. Ευχαριστώ, η κυρία Κατάινεν. Θα μιλήσω στη γλώσσα μου. Ευχαριστώ πολύ ε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πρώτα απ' όλα να πω ότι ε, συμφωνώ με τα όσα είπε η Μαρία Χίλθε προηγουμένως. Η συμφωνία αυτή αποτελεί τεράστιο επίτευγμα και είναι ιδιαίτερος ικανοποιητική γιατί δίνει πολλές ε, ευκαιρίες ας πούμε για τα γεωργικά προϊόντα. Πάνω από 80% των προϊόντων μας ε, θα διευκολυνθούν ε, στην διαμπόρευση τους μέσω αυτής της συμφωνίας. Επίσης, νομίζω ότι και η Ιαπωνική πλευρά έχει δεσμευτεί ισχυρότατα όσον αφορά το θέμα αυτό και αυτό είναι πολύ ικανοποιητικό. Αυτή η συμφωνία μας παρέχει πολλές ευκαιρίες ε, πρόσβασης στην ασιατική αγορά ε, και μάλιστα σε πολλούς και διάφορους τομείς. Ε, πρέπει επίσης να υπογραμμίσουμε, να προσέξουμε το γεγονός ότι εμείς ε, έχουμε ξεπεράσει τις Ηνωμένε Πολιτείε που μόλις τώρα ξεκινάει τέτοιες διαπραγματεύσεις. Ε, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όμως ε, υπέρ μας αυτό το προβάδισμα που έχουμε. Να ευχαριστώ λοιπόν, να ευχαριστήσω τον εισηγητή και την Κομισιόν. Ευχαριστώ η Μαρία Ρενά. Ευχαριστώ πολύ. Πράγματι, το ψήφισμα αποτέλεσε αντικείμενο διαφόρων τροπολογιών. Ήδη συζητήσαμε για κάποιες τροπολογίες οι οποίες έχουν κατατεθεί από μέλη της σοσιαλιστικής ε, ε, ομάδας. Ήθελα να ξέρω όμως ποιο είναι το καθεστώς αυτού του ψηφίσματος. Ε, είναι για να έχουμε καλή συνείδηση. Δεν είναι και πολύ καλό αυτό. Εάν στόχος του ψηφίσματος είναι να προχωρήσει κάποια στοιχεία αυτής της συμφωνίας, τότε καλό είναι να τη δουλέψουμε. Κατά την άποψή μου υπάρχουν τρεις σημαντικές προτεραιότητες. Πρώτο, το θέμα ε, των... Ε, ε των διαφωνιών όσον αφορά το Διεθνή Οργανισμό Εργασίας ε, μετά ε, ε, πιστεύω ότι έχουμε δει κάποια πρόοδο, όμως καμία διασφάλιση όσον αφορά την επικύρωση της συμφωνίας, της σύμβασης του Διεθνούς Οργανισμού εργασίας. Δεύτερον, ε, το να συζητούμε για ρήτρα αναθεώρησης ε, τη στιγμή που η ίδια η Κομισιόν μας είπε ότι δεν έχει καμία, ε, καμία διάθεση και πρόθεση να δουλέψει για μια ρήτρα βιώσιμης ανάπτυξης και με συγκεκριμένες κυρώσεις σε περίπτωση μη εφαρμογής, αυτό δεν μας δίνει καμία διασφάλιση. Εγώ θα ήθελα μέχρι να προταθεί κάτι πολύ συγκεκριμένο όσον αφορά την βιώσιμη ανάπτυξη και όχι μονάχα εργαλεία, τα οποία στην ουσία είναι εργαλεία διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών. Εγώ αναφέρομαι σε εργαλεία πολύ και μηχανισμούς πολύ πιο δεσμευτικούς όσον αφορά την βιώσιμη ανάπτυξη. Τρίτη προτεραιότητα, Συμφωνία των Παρισίων. Δεν νομίζω ότι η απλή αναφορά ε, της Συμφωνίας των Παρισίων συνεπάγεται και εφαρμογή της. Πρέπει να μιλήσουμε για συγκεκριμένα μέτρα όσον αφορά ε, την να την μείωση των ε, εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα ε, όσον αφορά την αποψήλωση των δασών. Μιλάμε για πράγματα για τα οποία η Ιαπωνία δεν έχει δείξει ακόμα συγκεκριμένα δείγματα γραφή ότι θέλει να προχωρήσει και επομένως λέω ότι οι απλές αναφορές και η ρήτρα αναθεώρησης δεν είναι αρκετά μέτρα. Ευχαριστώ. Κυρία Χάινς. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε υποβάλει και εμεί διάφορε τροπολογίε. Θέλουμε ένα δίκαιο εμπόριο. Σε ό,τι αφορά τι απαιτήσει, ε, σε ό,τι αφορά αυτό το κεφάλαιο με το μηχανισμό του κυρώσεων, για μας είναι σημαντικό. Ε, υπόθηκε ε, και εγώ δεν καταλαβαίνω πολύ καλά Το είχαμε δεχτεί την πρώτη φορά και το ΕΛΚ για τη Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία, Χιλή. Ε, το δέχτηκαν και το ΕΛΚ και άλλες ομάδες στα ψηφίσματα. Γιατί εδώ πρέπει να είναι διαφορετικά τα πράγματα. Επίσης, ε, αυτό το επιχείρημα δεν μπορούμε να τα πετήσουμε από την Ιαπωνία γιατί δεν θα μας εμπιστεύονται ή θα αποδυναμωθούν εμπορικές σχέσεις. Άμα μπορούμε να απαιτούμε κάτι, μπορεί να το απαιτεί και η Ιαπωνία, ε, αν υπάρχει αυτός ο μηχανισμός. Παραδείγματο χάρη, υπάρχουν ε, λόγω της ε, σοδιάς, της συγκομιδής, πολύ επισφαλής συνθήκες εργασίας και όλα αυτά πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας. Θέλουμε να βοηθήσουμε και να βελτιώσουμε την κατάσταση. Ό,τι αυτό το υπόλοιπο ε, του ψηφίσματος ε, είναι σαφές ότι πρέπει να αναφέρονται οι κανόνες ε, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και η επικύρωση των δύο συμβάσεων, συνθήκων που δεν έχει κυρώσει ακόμα. Το review clause επίσης πρέπει να αναφέρεται, αλλιώς δεν μπορούμε να ψηφίσουμε. Αν Μαρή Μινέρ. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον εισηγητή. Προσπάθησε να καλύψει διάφορες από τις ανησυχίες μας. Πολλά ακόμα παραμένουν, βέβαια. Ένα από τα προβλήματα είναι ότι η συμφωνία αυτή καλύπτει πολλά ζητήματα και είναι πολύ περίπλοκη. σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να δώσουμε λευκή επιταγή, να εξουσιοδοτήσουμε μια διαπραγμάτευση χωρίς περιορισμούς και αυτό φαίνεται και από τις πολλές τροπολογίες. Δεν επιθυμούμε τέτοιου τύπου συμφωνίες, οι οποίες τελικά δημιουργούν μια ενιαία αγορά με μεγάλες περιοχές του πλανήτη, χωρίς να έχουμε καμία διασφάλιση ότι εκείνες οι άλλες τρίτες χώρες ακολουθούν αντίστοιχα πρότυπα όσον αφορά το περιβάλλον και τους εργαζόμενους. Αυτά, αυτό του τύπου συμφωνίας είναι προς όφελος των πολυεθνικών εταιριών και όχι των πολιτών μας. Στη συμφωνία που συζητούμε δεν αναφέρονται σαφώς οι συμβάσεις του Παγκοσμίου Οργανισμού Εργασίας, ορισμένες από αυτές δεν τις έχει πυροκυρώσει η Ιαπωνία, και επίσης ακόμα και τα ζητήματα της βιώσιμης ανάπτυξης που αναφέρονται δεν είναι ξεκάθαρο πώς θα επιβάλλονται. Με ε, ενδιαφέρει επίσης ιδιαίτερα το ζήτημα της επισήμανσης των τροφίμων και της κατάστασης στην Ιαπωνία. Μπορεί να βρεθούμε με προϊόντα στην ευρωπαϊκή αγορά που δεν πληρούν τις δικές μας προδιαγραφές. Τέλος. Οποτεδήποτε προβλέπονται υποχρεώσεις, πρέπει να έχουμε και έναν μηχανισμό. Θα πρέπει λοιπόν να εισαχθεί στη συμφωνία και μια ρήτρα για ε, έναν μηχανισμό επίλυσης των διαφορών. Έχω υποβάλει σχετικές τροπολογίες. Ευχαριστώ. Κύριος Σιένφελτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πω ότι εάν, όπως ορισμένοι προτείνουν, το Κοινοβούλιο δεν δώσει τη σύμφωνη γνώμη του, και δεν επικυρωθεί αυτή η συμφωνία, τότε δεν βλέπω γιατί και πώς συμφωνήσαμε ε, με όλες τις προηγούμενες. Θα πρέπει να συγκρίνουμε τη συγκεκριμένη Συμφωνία Ελευθερού Εμπορίου με όλες τις προηγούμενες για τις οποίες το Κοινοβούλιο έχει δώσει τη Σύμφωνη του Γνώμη. Και ξεκάθαρα είναι η καλύτερη που έχουμε δει μέχρι τώρα. Ανταποκρίνεται στις ε, επιθυμίες μας, στις απαιτήσει μας, σε αυτό που θέλουμε να περιλαμβάνουν οι Συμφωνίες Ελευθερού Εμπορίου. Αναφέρεται για παράδειγμα σε ζητήματα βιώσιμη ανάπτυξη. Ο Χέλμου και άλλοι συνάδελφοι ε, είπαν τη δικιά τους θέση και πόσο αναφέ, ανησυχούν για τους εργαζομένους ή τους αγρότες στην ε, Ιαπωνία ή και συνολικά για την Ιαπωνική κοινωνία. Μάλιστα, τότε όμως θα σας προτρίνω να εξετάσετε τα στατιστικά στοιχεία για την κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη της Ιαπωνίας. Θα έλεγα ότι το 95% των χωρών του κόσμου θα ήθελα να βρίσκονται εκεί που βρίσκεται σήμερα η Ιαπωνία όσον αφορά την κοινωνικο-οικονομική τους ανάπτυξη ή σε οποιοδήποτε τομέα της ανάπτυξης ή της κατάστασης της κοινωνίας. Είναι μία από τις πλουσιότερες χώρες στον κόσμο στην Ευρώπη μιλώντας η Γερμανία είναι η πιο πλούσια χώρα και δεν καταλαβαίνω πώς οι Γερμανοί θα μπορούσαν να διαμαρτύρονται για το, το βιωτικό επίπεδο στη Γερμανία. Η Γερμανία είναι και αυτή μια χώρα η οποία στην παγκόσμια ιστορία δημιούργησε τεράστιους πολέμους με βαρύ φόρο αίματος. Γιατί το αναφέρω αυτό, γιατί και η Ιαπωνία είναι μια τέτοια χώρα. Είχαμε τον πόλεμο, τον βιώτατο φρικτό πόλεμο μεταξύ Κίνας και Ιαπωνίας. Γιατί τα λέω αυτά, γιατί υπάρχει μια αναλογία ανάμεσα σε αυτές τις δύο χώρες που είχαν ένα τέτοιο παρελθόν. Πώς κατάφεραν να το ξεπεράσουν με το να είναι ανοιχτές σε συνεργασία με άλλες χώρες, με άλλες περιοχές του πλανήτη. Με το εμπόριο και με την ανάπτυξη. Αυτό είναι καλό και βοηθάει τους εργαζόμενους, βοηθάει τους αγρότες, βοηθάει όλους τους ανθρώπους τους οποίους αναφέρετε. αναφέρατε. Οι άνθρωποι στο Τόκιο είναι ευτυχείς, επιθυμούν τη συμφωνία, τη σύναψη της συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσείς λέτε ότι θέλετε να τους προστατεύσετε και ανησυχείτε για αυτούς, εκείνοι την επιθυμούν. Thank you, Chair. First, I would like to... Ο κύριος Κάμπελικ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας για όλες τις προσπάθειες και επίσης γιατί κατέδειξε πόσο σημαντική είναι αυτή η συμφωνία και οικονομικά και στρατηγικά. Συμφωνώ και εγώ ότι αυτή η συμφωνία έχει μεγάλη αξία και πολιτική και οικονομική. Όχι μόνο θα αυξηθούν σημαντικά οι εξαγωγές, αλλά επίσης θα στείλει και ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να υποστηρίζει το ανοιχτό ελεύθερο εμπόριο με βάση κανόνες. Στη σημερινή εποχή με τον Τραμπ αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι ξεκάθαρο ότι και το εμπόριο και το ζήτημα της βιώσιμης ανάπτυξης είναι σημαντικά για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα και για αυτό να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Η Ιαπωνία είναι ένας κρίσιμος στρατηγικός εταίρο. Γι' αυτό είναι και συμβολικά πολύ σημαντικό ότι σε αυτήν τη συμφωνία με την Ιαπωνία έχουμε για πρώτη φορά μια αναφορά στην βιώσιμη ανάπτυξη και στη Συμφωνία των Παρισίων. το κεφάλαιο για την βιώσιμη ανάπτυξη από μόνο του θα είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έτσι ώστε να συνεχίσουν να συζητιούνται τα ζητήματα αυτά του περιβάλλοντος, του, των εργατικών δικαιωμάτων και επίσης των εκκρεμωτήτων με τις συμφωνίες του Παγκοσμίου Οργανισμού Εργασίας. Κύριε Πρόεδρε, παίρνω το λόγο ως σκιώδης εισηγητής ε, για να απαντήσω σε ένα ε, σχόλιο των, ε, της συγκεκριμένα της συναδέλφου της Σοσιαλίστριας από το Ηνωμένο Βασίλειο. Είπαμε ότι έχουμε ψηφίσει επανειλημμένα λέμε, αλλά αναφερόμαστε στο κείμενο για την Αυστραλία και την Νέα Ζηλανδία και παραθέτω το ενδεχόμενο να υπάρχει υπάρξουν κυρώσεις. Αυτό δεν σημαίνει επιβολή κυρώσεων άμεσα. Επίσης, η κυρία Αρενά μας είπε ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ε, εφαρμογή των δύο συμβάσεων του Διεθνούς Οργανισμού ε, Εργασίας Πρόκειται για ένα ζήτημα όντως το οποίο δεν απαντήθηκε καθαρά. Εμείς πιέσαμε στις ε, ε επαφές μας και στις συνεδριάσεις ε, και ε, έχουμε και μία επιστολή του πρέσβεως Κουνταμά ε, όπου σαφώς αναφέρει ότι η κυβέρνηση της Ιαπωνίας αποφάσισε ε, να ε, οργανώσει την πρώτη συνεδρίαση μεταξύ Υπουργών τον μήνα Οκτώβριο έτσι ώστε να δει με ποιο τρόπο κλπ. Η Ιαπωνία θα υλοποιήσει κλπ. Κατά την άποψή μου αυτή είναι μια σαφής διατύπωση και επομένως πιστεύω ότι, Η, ε, ότι μπορεί κανείς να έχει αρκετή εμπιστοσύνη ότι τα πράγματα θα προχωρήσουν καλά και είμαι ε, ε, βέβαιος ότι θα βρούμε και ε, αν έχετε κι εσείς καλή θέληση θα βρούμε οπωσδήποτε μια διατύπωση που να μας αρέσει σε όλους. Πάρα πολύ ωραία λέει ο Πρόεδρος, είναι πολύ ωραία που έχουμε τόσο ζωντανή συζήτηση σε τούτη την Επιτροπή. Αυτό πραγματικά μας δίνει κέφι και θέλουμε να συζητούμε. Θα δώσω τώρα το λόγο στην Επιτροπή, στον κύριο Μάρκο Σιρόλο έτσι ώστε να συμβάλλει και αυτός σε αυτή τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Πρώτα απ' όλα η Κομισιόν θα ήθελε να ευχαριστήσει τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πήραν το λόγο σε αυτήν την ενδιαφέρουσα συζήτηση επί μιας πολύ σημαντικής συμφωνίας. Θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια επί τη βάση των όσων ε, ακούσαμε για να δώσω και εγώ τη δικιά μου συμβολή στη συζήτηση. Πρώτον, αναφέρθηκε από πολλούς βουλευτές ότι είναι μεγάλη αξίας, στρατηγικής αξίας αυτή η συμφωνία διότι πραγματικά ενισχύει τις σχέσεις με έναν εταίρο με τον οποίο ε, ε, ε, μοιραζόμαστε κοινέ αξίες και κοινά πρότυπα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί οι καιροί είναι δύσκολοι και είναι σημαντικό να έχουμε μία τόσο στρατηγική εταιρική σχέση με έναν πολύ ισχυρό στενό φίλο και έναν επιφανή εταίρο στη διεθνή σκηνή. Το θέμα των αξιών και των προτύπων επίσης είναι πολύ σημαντικό. Άκουσα κάποια μέλη ε, να αναφέρονται στον κίνδυνο, τον ενδεχόμενο κίνδυνο μείωσης ε, των ε, προτύπων Πραγματικά δεν διατρέχουμε κανένα κίνδυνο ε, μείωση των προτύπων όσον αφορά την ασφάλεια και την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων, γιατί πραγματικά όσον αφορά την προστασία του καταναλωτού και την προστασία των τροφίμων, ε, ε, τα πρότυπα είναι εξαιρετικά υψηλά εις την Ιαπωνία. Επίσης πιστεύουμε ότι θα υπάρξει άμεσα ε, απόλυτη ισοτιμία των εξαγωγών, των εξαγωγών μας και των εξαγωγικών εταιριών ε, προς την ε, Ιαπωνία άμεσα μετά την ισχύ της συμφωνίας όσον αφορά το κρασί, ναι και εδώ θα βρισκόμαστε σε ίδιο επίπεδο με άλλους παραγωγούς. Uh, uh, in this uh, ε, και με άλλους ε, παίκτες για παρόμοια ε, προϊόντα. Επίσης, όσον αφορά το DST, νομίζω ότι είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε, όπως άλλωστε έγινε, την επιστολή, να υπενθυμίσουμε λέω την επιστολή του πρέσβεως Κουντάμα, είναι σημαντική η επιστολή αυτή και το περιεχόμενό της, γιατί πρόκειται για μία, ε, ε, για μία επίσημη επιστολή ενός απολύτου πληρεξουσίου και εντολοδόχου της ε, ε κυβέρνησης της Ιαπωνίας, όπου γραπτά πλέον αναφέρεται στο θέμα αυτό και οπωσδήποτε θα ακολουθήσει επίσημη θέση από το Τόκιο. Ε, είναι μια πολύ καλή αρχή, είναι μια πολύ καλή κίνηση ε, και επομένως ε, περιμένουμε τα καλύτερα, διότι με τον τρόπο αυτό αυξάνεται και το δυναμικό της στενής μας συνεργασίας και για το θέμα αυτό. Ε, επίσης για τη Συμφωνία των Παρισίων ε, είπατε ότι ε, απλώς γίνεται αναφορά. Όχι, πρόκειται για δέσμευση, γιατί στα αγγλικά λέγεται ότι the parties shall. Επομένως είναι κάτι υποχρεωτικό, είναι κάτι δεσμευτικό. Επίσης όσον αφορά την παράνομη ξυλία και την παράνομη υλοτομία εδώ και ένα χρόνο έχει αρχίσει ε, να ε, υλοποιείται η συμφωνία ε, και πραγματικά να σας πω ότι από την 19η Σεπτεμβρίου υπάρχει πλέον ένας κατάλογος των καταχωρισμένων εταιριών οι οποίες έχουν, είναι μέσα στο πρόγραμμα το αναγνωρισμένο ας πούμε. Πρόκειται για 39 εταιρείες οι οποίες έχουν δεσμευτεί να προχωρήσουν, να προωθήσουν αυτό το εργαλείο ως ένα εργαλείο ε, ε, που σηματοδοτεί την υπευθυνότητα των εμπλεκομένων. Βεβαίως συνεχίζουμε στενή συνεργασία με την Ιαπωνία και η οδός που έχει ξεκινήσει και η κατεύθυνση που παίρνει η κατάσταση είναι πολλά υποσχόμενη. Η τελευταίο σχόλιο, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, ε, έγινε μια αναφορή, αναφορά σχετικά με το γεγονός ότι θα μπορούσε να ανοίξει η πόρτα για μεγαλύτερη κρίση. Ε, το κεφάλαιο των υπηρεσιών, κυρίως δεν των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, προσπαθεί να μειώσει, βλέπε να καταργήσει ε, ορισμένα προσκόμματα, αλλά από την άλλη πλευρά... Παρόλα αυτά, δίνει την δυνατότητα να ληφθούν προληπτικά μέτρα. Δεν καταλαβαίνουμε λοιπόν πού ε, έγκυται ο κίνδυνος ε, στο κεφάλαιο των υπηρεσιών. Απλώς διασφαλίζεται ότι οι δικοί μας εμπορευόμενοι θα έχουν την δυνατότητα να παρέχουν υπηρεσίες τις οποίες έχουν την αδειοδότηση να παρέχουν ή ε, εσωτερική πάροχοι. Ε, επί τη βάση της γενικής αρχής ε, της μη διακριτικής μεταχείρισης. Αυτή η αρχή άλλωστε της μη διάκρισης ε, δεν αφορά μονάχα το κεφάλαιο των υπηρεσιών, αλλά και άλλα κεφάλαια, επομένως δεν κατανοώ που υπάρχει ο κίνδυνος. Αυτά τα ολίγα και σας ευχαριστώ. Κύριος Μάρτιν, ήταν πολύ σύντομος. Ξέρω τις απόψεις του Πέδρο, ουσιαστικά εκ θα καταλήξω για το ερώτημα της Μαρία Ρενά. Θέλουμε απλά ε, να κοιμούμαστε τον ύπνο του δικαίου ε, ή θέλουμε να αλλάξουμε συμφωνία με το ψήφισμα. Όχι, εμείς θέλουμε, ε, ο εισηγητής τουλάχιστον, ε, να Λέμε στο ψήφισμα ότι η επικύρωση θα πρέπει να γίνει το σύντομα των δυνατόν και θέλουμε να συνεχίσουμε να σκούμε πιέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιαπωνία για να τηρήσουν τι δεσμεύσει του σε ό,τι αφορά ε, την ξυλία, τη Συμφωνία των Παρισιών και όλε τι διατάξει. Ε, ε μεγάλη σημασία στο κεφάλαιο εμπορίου βιώσιμη ανάπτυξη κτλ. Ένα άλλο σχόλιο που θέλω να κάνω προς τον Άνταμ, τον οποίο εν γίνει συμφωνώ, αλλά σε μια εμπορική συμφωνία υπάρχουν οι και οι τιμένοι και οι τιμένοι θα υπάρξουν από την εμπορική συμφωνία. Ίσως οι Ιαπωνέζοι οι μικροί αγρότες ε, να πληγούν. Πρέπει να είμαστε ειλικρινεί. Αυτή είναι, είναι λυπηρό βέβαια, αλλά αυτή είναι η κατάληξη. Κάποιοι από μια εμπορική συμφωνία θα κερδίσουν, κάποιοι θα χάσουν ω ε, Συμβούλιο και, ω Επιτροπή ε, θέλουμε να φροντίσουμε το κύριο να είναι πολύ περισσότερο των ζημιών, των απολειών που πιστεύω ότι έτσι θα ισχύει και θα δημιουργηθεί ένα καλύτερο περιβάλλον και συνθήκες ε, θετικές ε, στο εμπόριο, το παγκόσμιο και αυτό είναι θετικό. Ευχαριστώ πρόεδρο. Εδώ ολοκληρώνουμε λοιπόν τη συζήτηση των τροπολογιών του ψηφίσματος ε, για την Ιαπωνία και τώρα θα περάσουμε στο σημείο 6 που είναι η εμπορική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, Περού και Κολομβίας. Συγητής ο κύριος Φίσας. Πριν του δώσω το λόγο, θέλω να καλωσορίσω τον Υφυπουργό Εμπορίου του Περού, τον κύριο Έντγκαρ Βάσκες και τον πρέσβη της Κολομβίας, Φρανσίσκο Κόι Γρανάδος. Κύριε Φίσας, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, και τον και τους πρέσβεις για την παρουσία τους. Η συμφωνία με την Κολομβία και το Περού ε, επί πέντε χρόνια ε, ε, εφαρμόστηκε de este informe que presentamos Προσωρινά. Ε, και ε, βεβαίως πρέπει να πούμε ότι ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η επιτήρηση των εμπορικών συμφωνιών αποτελεί δικαιοδοσία του Κοινοβουλίου και υποχρέωσή του και στη διάρκεια της συμφωνίας και στη διάρκεια της υλοποίησης. Βεβαίως εδώ μιλάμε για εμπορικές συμφωνίες οι οποίες όμως βασίζονται σε κοινά πρότυπα, κοινέ αξίες και γενικώ στοιχεία τα οποία μπορούν να έχουν θετικό αντίκτυπο στον κοινωνικο-οικονομικό ε, ε, χαρακτήρα και στην κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη των χωρών. Είναι πολύ σημαντική σε σημασία σε αυτή ε, η συμφωνία γιατί η Λατινική Αμερική είναι σημαντικός εταίρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι γεγονός ότι η διμερή, το διμερές εμπόριο λόγω και της συγκυρίας δεν έχει αναπτυχθεί αναπτυχθεί ωστόσο έχουν έχουν αντισταθμιστεί οι αρνητικές ροές. Σταθεροποιήθηκε, βελτίωσε την σταθεροποίηση, την οικονομική κατάσταση στο Περού και την Κολομβία. Είναι σημαντικό για τις χώρες αυτές να έχουν ε, κάποιο, ε, ε, κάποια αγορά αναφορά εκτός της Λατινικής Αμερικής. Μέσω της συμφωνίας η Κολομβία και το Περού διαφοροποίησαν και εμπλούτησαν τις εξαγωγές τους με πολύ, καλές, πολύ καλό αντίκτυπο για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις τους. Όσον αφορά τώρα την, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, της ευρωπαϊκής ε, πλευράς, ε, η συμφωνία αυτή σήμαινε άρση των διμερών εμπορικών φραγμών και βελτίωση των εμπορικών ροών. Επίσης, οι μικρομεσαίες μας επιχειρήσεις πρέπει να πούμε ότι πολύ συχνά δεν γνωρίζουν τις, τις δυνατότητες που, δίνουν αυτές, που δίνει αυτή η συμφωνία και επομένω και τα κράτη-μέλη και η Κομισιόν θα πρέπει να πράξει τα δέοντα έτσι ώστε να μπορέσουν και οι δικές μας επιχειρήσεις ε, να ε, ε, απολαύσουν των πλέον εκτιμάτων που παρέχει αυτή η <clears throat> συμφωνία. Ε, όσον αφορά φυ... Ε, υγειονομικά και φυτοϊγειονομικά θέματα παραμένουν κάποια ζητήματα ε, όπως ε, ε η πιστοποίηση κάποιων προϊόντων κρέατος και γαλακτοκομικών. Επίσης οι φόροι που μπορούν να εφαρμοστούν σε εισαγόμενα τρόφιμα. Επίσης είναι δύσκολο για ε, την Κολομβία και το Περού να ε, ε, συμφωνήσουν με κάποιες και να εφαρμόσουν μάλλον κάποιες κάποια πρότυπα και να συμμορφωθούν με τα πρότυπα αυτά όσον αφορά γεωγραφικές ενδείξεις κλπ. Στόχος πρέπει να είναι η κοινή εργασία έτσι ώστε τα οι διεθνείς συμφωνίες για τα εργασιακά να εφαρμοστούν σωστά. Έχουν γίνει προσπάθειες από πλευράς Κολομβίας και Περού, αλλά ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Ε, ε πρέπει να συνεχίσει η υλοποίηση του οδικού χάρτη ε, όσον αφορά τις ε, ε που αφορούν τα εργασιακά δικαιώματα, το περιβάλλον, την εργασία ε, των ανηλίκων, την, το δικαίωμα του συνεταιρίζεστε κτλ. Ε, μας ε, ενδιαφέρει επίσης το κεφάλαιο της βιώσιμης ανάπτυξης και η υλοποίηση ε, των αρχών αυτών και χαίρομαι που είναι εδώ ο κύριος Υπουργό, έτσι ώστε να ακούσω και τη δικιά του άποψη για τα θέματα αυτά. Ένα άλλο σημείο το οποίο αναφέρω στο κείμενό μου είναι η δυνατότητα της κοινωνίας των πολιτών του, της Κολομβίας και του Περού ε, να μπορέσουν ε, μέσω των συμβουλευτικών ομάδων, των advisory groups, να συμμετάσχουν πλήρως στην συμφωνία. Ε, και σημαντικό είναι, και αυτό θα δώσει και προστιθέμενη αξία, να είναι ανεξάρτητες. Γι' αυτό λοιπόν χαίρομαι που η Κολομβία έχει εφαρμόσει τέτοιες ομάδες και θα έπρεπε και το Περού το ενθαρρύνω να κάνει το ίδιο. Είναι γεγονός ότι ε, δεν είναι ίδια η κατάσταση στην Κολομβία και στον Περού με την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε αυτές τις φίλες χώρες ε, να προχωρήσουν στον δρόμο αυτό της συμμόρφωσης των προτύπων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης το γεγονός της προσχώρησης της Κολομβίας στον ΩΣΑ στις 30 Μαΐου του 2018 και ενθαρρύνω την, το Περού να συνεχίσει προς την ίδια κατεύθυνση κατεύθυνση. Ε, σας διαβεβαιώ ότι είμαι ανοιχτό για την καλή συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων έτσι ώστε εν τέλει το κείμενο του Κοινοβουλίου να είναι ε, σωστό. Ευχαριστώ. Για τους σοσιαλιστές, ε, δύο λεπτά. Η Μακουλάδα. Πρώτα απ' όλα να καλωσορίσω τους εκπροσώπους της κυβέρνησης ε, και της πρεσβείας από το Πέρο και την Κολομβία και να συγχαρώ τον εισηγητή για την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει, για την πολύ καλή έκθεση που μας παρουσίασε ως βάση και σας λέω ότι πιστεύω πως ε, μέσω της συνεργασίας μεταξύ εισηγητούς και οδών και μέσω της κατάστροπολογιών σίγουρα θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία που θα την υποστηρίξει μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη πλειοψηφία. Σε ό,τι αφορά τα εμπορικά αποτελέσματα, τη διαφοροποίηση των εξαγωγών, βλέπουμε θετικά αποτελέσματα και για την περίπτωση της και την περίπτωση του Πέρου. Επίσης, η συμφωνία αυτή έχει στρατηγική σημασία γιατί θα βοηθήσει σε ε, ιδιαίτερες καταστάσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες ε, για να ε, απαλληλθούν τα σημεία τριβής και οι αντιπαραθέσεις που μπορεί να υπάρχουν και να προωθηθεί βιώσιμη ανάπτυξη. Προκλήσεις παραμένουν, αυτό είναι αλήθεια, όπως αλήθεια είναι ότι κατά την άποψή μας σημαντικό είναι να υπάρξει πλήρης προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων η διακριτική φορολόγηση των πνευματοδών που εισάγονται επίσης είναι ένα θέμα και κάτι πάρα πολύ σημαντικό για το Κοινοβούλιο και ιδίω για την ομάδα που εκπροσωπώ είναι η τήρηση του δικού χάρτη σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα, κοινωνικά δικαιώματα και εργασιακά δικαιώματα και σε ό,τι αφορά το κεφάλαιο βιώσιμη ανάπτυξη. Πολλές φορές εδώ στην Επιτροπή μας Έχουμε πει ότι είναι σημαντικό να υπογράφεται μια καλή συμφωνία, αλλά εξίσου σημαντικό να εφαρμόζεται πλήρω. Υπάρχουν πτυχέ τι οποίε χρειάζεται χρόνο μέχρι να μπορέσουν να εφαρμοστούν, αλήθεια είναι και αυτό. Όμω πρέπει να υπάρχει πολύ πιο επικαιροποιημένη ενημέρωση με δείκτε ε, για να βλέπουμε τι κάνουν και δύο χώρε. Πώς εφαρμόζουν το κεφάλαιο της βιώσιμης ανάπτυξης. Το Κοινοβούλιο οφείλει να, μάλλον πρέπει να ενημερώνεται πολύ περισσότερο σε ό,τι αφορά ιδίω αυτό το κεφάλαιο και την εφαρμογή του. Ζητώ λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας δίνει και μας ενημέρωση ε, και το ζητώ και από τις αρχές της Κολομβίας και του Πέρου. Ένα άλλο στοιχείο σημαντικό είναι η διάρθρωση του διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών, το είπε και παίρνουμε καταγγελίες από την κοινωνία των πολιτών και πήγαμε με επίσημη αντιπροσωπεία και το επιβεβαιώσαμε επιτόπου. Άρα πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερες προσπάθειες και από τις δύο πλευρές και ιδίω από την κυβέρνηση του Περού ώστε να υπάρξει δομημένος διάλογος και εκπροσώπηση της κοινωνίας των πολιτών. Θα καταθέσουν τροπολογίες για να βελτιώσουμε ορισμένες πτυχές του κειμένου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Ζαραντήλη από το ECR, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κύριο Φίσας για μια αναλυτική και επικοδομητική έκθεση τις οποίες μπορεί να βασιστεί η συζήτηση στην Επιτροπή μας. Σε μεγάλο βαθμό συμφωνώ. Θα ήθελα να επισημάνω το εξής πρέπει να γνωρίζουμε τον αντίκτυπο αυτής της ε, συμφωνίας. Το αναφέρει και στο σημείο 10. Πολλές από τις μικρομεσές επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν γνωρίζουν ότι έχουν δυνατότητες καινούριε που τους έχει δημιουργήσει αυτή η συμφωνία. Φαίνεται αυτό πράγματι. Ε, η Κολομβία και το Περού ήταν εκείνοι οι οποίοι κέρδισαν περισσότερο, θα έλεγα περισσότερο από αυτή τη συμφωνία. Ακόμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουμε δει τα ωφέλη. Έχουμε ένα έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου που όχι μόνο δεν έχει μειωθεί, αλλά έχει αυξηθεί κατά 14% από το 2017. Επομένως, το ερώτημα είναι τι μπορούμε να κάνουμε συγκεκριμένα για να υπάρξει μεγαλύτερη ε, ευαισθητοποίηση, γνώση των επιχειρήσεων για τις ευκαιρίες που τους δίνει αυτή η συμφωνία. Θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις του εισηγητή μας, ειδικά για αυτό το θέμα. Το δεύτερο, που ήθελα να επισημάνω είναι το ζήτημα της διαφθοράς. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι, είναι κάτι το οποίο μας το αναφέρουν και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, διαμαρτύρονται γι' αυτό. Και πρέπει να δούμε τι έχει αλλάξει από τότε που συνήφθη η συμφωνία και επίσης τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε ε, με μέτρα καταπολέμησης της διαφθοράς. Και τρίτον και τελευταίο, κοιτώντα το ζήτημα γενικότερα γεωπολιτικά, και θα εστιαστώ περισσότερο στο Περού εδώ, μιας και είναι από τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, μια από τις χώρες που υποστηρίζει περισσότερο το ελεύθερο εμπόριο. Και έχοντα υπόψη και τις διαπραγματεύσεις για την TTIP, καλό θα ήταν να μας κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια ανάλυση για το πώς διεξήχθησαν οι διαπραγματεύσει που ε, ε, πώς προσέγγισε τις διαπραγματεύσεις ε, συγκρίνοντας την TTIP και αυτή τη συμφωνία, ιδίως για τα ζητήματα του περιβάλλοντος και κατά τα άλλα είμαστε έτοιμοι να έχουμε μια επικοδομητική συνεργασία με τον εισηγητή. Σας ευχαριστώ κυρία Χίρς από την Άλτε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, αξιότιμοι εκπρόσωποι του Περού και της Κολομβίας, υποστηρίζουμε και εμείς την έκθεση, θεωρούμε ότι είναι πληρότατη. Ε, φαίνεται ότι οι συμφωνίες με το Περού, με την Κολομβία, τώρα πια και με τον Ισημερινό, είχαν πολλά θετικά αποτελέσματα. είχαμε ουσιαστική προόδο. Ζητήματα τα οποία κρεμούν ακόμα είναι το ζήτημα της δικαιοσύνης, της καταπολέμησης της διαφθοράς. Όμως... Είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, ό,τι αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις χώρες της Νότιας Αμερικής, ε, θέλουμε και αυτές να ωφεληθούν και είναι πολύ καλό. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι χρειάζονται περισσότερες ευκνήσεις εδώ και ενημέρωση και στην Ευρώπη για να μπορέσει να υπάρξει εκμετάλλευση αυτής της ευκαιρίας. Και θέλουμε να τονίσουμε ότι στην Κολομβία έχει, ε, υπάρχει ανάγκη να ξεκινήσει μια διαδικασία για να υπάρξει σταθερότητα για τις επενδύσεις, ε, για τη ε, δημιουργία εταιρικών σχέσεων στον κοινωνικό τομέα και εκεί που χρειάζεται, θεωρώ, κάποια αλλαγή είναι ο διάλογος με την κοινότητα των πολιτών. Und, ähm, es ist wichtig, dass wir hier... Είναι πάρα πολύ γρήγορο. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, να ε, υπάρξει ε, συνεργασία με τη νέα ε, κυβέρνηση της Κολομβίας και να μπορέσουμε να συνεργαστούμε εμάς, ε, για εμάς φιλελεύθερους. Είναι σημαντικό. Καταθέσουμε λοιπόν τροπολογίες ε, και τη ψηφιακή οικονομία για την Νότια Αμερική αλλά και την Ευρώπη. Θέλουμε να τονίσουμε τη σημασία της ψηφιακής οικονομίας. Θα καταθέσουμε σχετικές τροπολογίες και γι' αυτό ως φιλελεύθεροι ε, θεωρούμε ότι η σταδική αυτή εταιρική σχέση έχει μεγάλο δυναμικό και είναι καλή η κατεύθυνση που έχουμε ακολουθήσει. Ευχαριστώ πολύ. Ο Χέλμουντ Σόλτ εκ μέρου τη ΓΚΟΕ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγητή για την εξαιρετικά αναλυτική έκθεσή του. Κάτι που κατά την άποψή μου είναι σημαντικό. Προσπαθούμε να αξιολογήσουμε μια πενταετή προκαταρκτική εφαρμογή της συμφωνίας. Εκκρεμεί ακόμα η επικύρωσή της από δύο κρατημέλη. Επομένω, δεν είναι μυστικό ότι αυτή η συμφωνία ήταν μια από τις συμφωνίες σε οποία δημιούργησε τις περισσότερες διαφωνίες και συζητήσεις. Γιατί πρόκειται για δύο χώρες με ιδιαιτερότητες Μιλώντας για την Κολομβία είχαμε τον εμφύλιο πόλεμο που καθόρισε ουσιαστικά τη συζήτηση για το ποια θα πρέπει να είναι η σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη χώρα αυτή. Και τώρα και στο μέλλον. έτσι ώστε η συνεργασία οικονομική, η πολιτική να είναι προς όφελος των πολιτών. Κάτι αντίστοιχο είχαμε και με το Περού. Ε, ε ήταν επίλυση αυτών των ζητημάτων ήταν προϋπόθεση που είχε θέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο πριν πέντε χρόνια. Και θα έλεγα ότι αυτή η συμφωνία είναι ένα από τα πιο συγκεκριμένα εργαλεία που έχουμε. Χρειάζεται λοιπόν μια εξέταση δίπλευρη που το λέει, λέει και η έκθεση αυτό. Δεν μπορούμε να πούμε ότι υπήρξαν και ε, βελτιώσεις αλλά και προβλήματα που συνεχίσουν να υπάρχουν. υπάρχουν. Πώς μπορούμε να συνεχίσουμε αυτή τη διαδικασία με τρόπο επικοδομητικό. Ε, ε, ε, έχουμε μπροστά μας τις εργασίες της ομάδας για την ολοκλήρωση της συμφωνίας και έχουμε επίσης και τις συμβουλευτικές ομάδες στο εθνικό επίπεδο. Το ερώτημα είναι πόσο αυτές είναι αντιπροσωπευτικές. Δυστυχώς, διαπιστώνουμε ότι στο εθνικό τοπικό επίπεδο υπήρξε μεγάλη υπονόμευση, καταστροφή και, ε, και, και, Γνωρίζουμε ότι έχουμε μία ε, δολοφονία κάθε δύο μέρες. Ε, αυτό δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε. Πρέπει να το συζητήσουμε και χαίρομαι που είναι παρόν και ο Υφυπουργό και οι πρέσβεις. Αλλά ε, πρέπει να συζητηθεί αυτό το συζήτημα και με τη συνεργασία μη κυβερνητικών οργανώσεων που μπορεί να μας δώσουν πληροφορίες για το πώς λειτουργούν τα πράγματα αυτές στις χώρες αυτές. Η κυρία Κιόρτον Ντάρλινγκ. Ευχαριστώ. Θα συνεχίσω από το ζήτημα που έθεσε ο Χέλμοντ. Όταν επικυρώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η συμφωνία αυτή πριν τι προηγούμενε ευρωεκλογέ, ήμουν τότε στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία. Και προσπαθούσαμε να θέσουμε το ζήτημα της βελτίωσης της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων στην Κολομβία και το Περού. Γι' αυτό λοιπόν κατά μία έννοια είναι θετικό, κατά μία έννοια είναι απογοητευτικό να βλέπει κανείς τις εξελιξείς. Διαπιστώνουμε πρόοδο στις διμερείς σχέσεις τις εμπορικές, όμως αυτό που κατά την άποψή μου λείπει από την έκθεση του εισηγητή και θα υποβάλω σχετικές τροπολογίες, είναι μια αναφορά και μια περιγραφή της κατάστασης επιτόπου, που το ανέφερε ο Χέλμοντ. Οι δολοφονίες, των αντιφρονούντων, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κολομβία. Ακόμα και μετά και ιδιαίτερα μετά τη συμφωνία ε, για τη λήξη του εμφυλίου. Δεν υπάρχει κάποια τέτοια αναφορά στην έκθεση, ούτε αναφέρεται επίσης η σχέση μεταξύ της προστασίας του περιβάλλοντος και των συγκρούσεων για την ιδιοκτησία της γης που έχουν οδηγήσει σε δολοφονίες ε, υπηρεσιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ηγετών κοινωνικών ομάδων στις χώρες αυτές. Πρέπει να αναφερθούμε σε αυτά. Επίσης πρέπει να αναφέρουμε ότι σε μεγάλο βαθμό οι εξαγωγές από αυτές τις δύο τις χώρες σχετίζονται με τους φυσικούς τους πόρους. Εάν λοιπόν μας ενδιαφέρει ουσιαστικά η τήρηση του οδικό χάρτη πρέπει να αναφερθούμε και σε αυτό. Στην Κολομβία επίσης έχουμε το υψηλότερο ποσοστό φόνων και εκφοβισμού συνδικαλιστικών ηγετών. Μόνο στο πρώτο εξάμεινο, μέχρι τον Αύγουστο μάλλον του 2018, 40 συνδικαλιστές δολοφονήθηκαν στην Κολομβία. από το 2012 στο 2017 έχουμε 217 παραβιάσεις του δικαιώματος στη ζωή, στην αξιοπρέπεια και στην ελευθερία της έκφρασης συνδικαλιστικών ηγετών με βάση εκθέσεις ε, αξιόπιστων διεθνών μη κυβερνητικών οργανώσεων και όλα αυτά δεν αναφέρονται στις εκθέσεις. Πιστεύω ότι πρέπει να αναφερθούμε στην πραγματικότητα ε, στο πεδίο, επιτόπου. Γιατί διαφορετικά δεν μπορούμε να έχουμε μια θετική επίδραση στην κατάσταση στις χώρες αυτές. Σας ευχαριστώ κυρία Αρένα. Σύντομα, συμφωνώ με αυτά που είπε η Τσούτ και θα ήθελα η έκθεση αυτή να εγγραφεί στο πλαίσιο του αποτελέσματος των εκλογών για την Κολομβία μιλάω, όπου η κυβέρνηση δεν έχει οδικό χάρτη για την εφαρμογή της Ειρηνευτικής Συμφωνίας. Ο κ. Ντούκε ήταν ε, κατά της Ειρηνευτικής Συμφωνίας στην προεκλογική του εξαρτία και θα ήταν ενδιαφέρον να σχετίσουμε την εφαρμογή της Ειρηνευτικής Συμφωνίας και του οδικού χάρτη με ε, την εμπορική συμφωνία, στον βαθμό που έχουμε και την πρόσβαση στη γη, την ιδιοκτησία. Και όπως είπε και η Τζούντ, εγκλήματα κατά υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ξέρουμε ότι γίνονται έχουν σχέση με παράνομη αλλά και νόμιμη εξωτερική δραστηριότητα, εφαρμογή της Ειρηνευτικής Συμφωνίας. Άρα, καλό είναι στο ψήφισμα να μπορέσουμε να βάλουμε αυτό το σημείο. Η Ευρώπη πολύ δραστήρια στήριξε όχι τη διάδικαση αλλά την Ειρηνευτική Συμφωνία αυτή καθ' αυτή και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το ε, αναφέρουμε. Στόχο τη εμπορική συμφωνία είναι η στήριξη μια τέτοια διαδικασία. Δεν μπορεί λοιπόν απλά η να ε, περιοριστεί στι εμπορικέ συναλλαγέ, αλλά και υπό το πρίσμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε μια χώρα όπω η Κολομβία σήμερα. Ευχαριστώ. Η Κάρολιν Γκράσφαντερ Χάιντ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ θέλω να μιλήσω για πράγματα που δεν είναι τόσο θετικά. Σίγουρα ε, κάποια πράγματα κινούνται προ σωστή κατεύθυνση, αλλά θα πρέπει να είμαστε ειλικρινεί και ανοιχτοί και να πούμε ότι πολλά δεν εφαρμόζονται. Και αυτό το οποίο με ανησυχεί ιδιαίτερα είναι τι γίνεται με του ε, αυτόχθονε ή με τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, όπω αναφέρθηκε, ή οι υπερασπιστέ δικαιωμάτων που διώκονται, που δολοφονούνται, όπω και συνδικαλιστέ. Το κεφάλαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων λοιπόν είναι πάρα πολύ αδύναμο και πρέπει να ενισχυθεί. Επίση, ό,τι αφορά τη συμμετοχή τη κοινωνία των πολιτών, συνέχεια ακούμε ότι υπάρχει πρόβλημα, πρέπει να υπάρξει ενίσχυση, πρέπει να συμμετάσχουν περισσότερο και εκεί νομίζω ότι πρέπει ε, να πιέσουμε περισσότερο. Επίσης αν υπάρχει παραβίαση, ε, τι θα γίνει με την ε, συμφωνία. Δεν μπορούμε να διαπραγματευόμαστε και να έχουμε θετική έκφαση αν δεν μπορούμε να ε, έχουμε κάποια μέτρα σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι διατάξεις και γι' αυτό θα καταθέσουμε τραπολιστικές. Κύριε Γιώργεν, Σερματίας Γιώργεν, σε Κομισιόν, τι λέει, έχετε τρία λεπτά στη διάθεσή σας. Uh, σας ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ κατάλληλη χρονική στιγμή κατά την οποία προσφέρεται ε, η, παρουσίαση της εκθεσής σας, γιατί είμαστε στο, είμαστε στο μέσον μάλλον αυτής της εφαρμογής. Έγινε μεγάλη πρόοδος τα τελευταία πέντε χρόνια. Βέβαια παραμένουν ακόμα πολλά άλλα που πρέπει να γίνουν, ιδίω το ζήτημα της πρόσβασης στην αγορά, το, της υφαντουργίας, ε, το ζητήματα στην Κολομβία ε, Έχουμε ζητήματα, για παράδειγμα, σε σχέση με τις δημόσιες προμήθειες, ε, δημόσιες συμβάσεις, ε, πρόσφατε αποφάσει που πρέπει να εφαρμοστούν. Επίση πρέπει να υπάρξει πρόοδο στον τομέα τη ε, βιώσιμη ανάπτυξη και τη σχέση του με το εμπόριο. Εδώ θεωρούμε ότι έχουν γίνει κάποια θετικά βήματα, αλλά πρέπει να αναλυφθούν πρωτοβουλίε και από τη δική μα πλευρά, αλλά σίγουρα και από την πλευρά των εταίρων μας της Άνδης, ιδιαίτερα το Περού. Ξεκινάει επίσης και η συνεργασία με τον Ισημερινό. Από εκεί, από την πλευρά της Κολομβίας, έχουμε δει κάποια ενθαρρυντικά βήματα. Έχουν δημιουργήσει κάποιες δομές οι οποίες είναι απαραίτητες για να συμμετέχει η κοινωνία των πολιτών. Παρατηρούμε λοιπόν ακούμε και θα εξετάσουμε εις βάθος αυτά που αναφέρει η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ξεκινήσουμε και εμείς μια εις βάθος αξιολόγηση αντικτύπου προς το τέλος της χρονιάς. Και βέβαια υπάρχει και το ζήτημα του της ε, δημιουργίας του μηχανισμού επίλυσης συγκρούσεων που θα πρέπει να ε, δημιουργήσουμε ε, σε συνεργασία με αυτές τις δύο χώρες. Σας ευχαριστούμε για την έκθεσή σας. Σας ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στον, στην, στον Υφυπουργό, όχι, συγγνώμη, συγγνώμη, ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Και... Ζαν Πιεμπό, έχετε το λόγο. Αναπληρωτής ήταν ο αναπληρωτηματάρχης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να σας ευχαριστήσω που μου δώσετε την ευκαιρία και εμένα να σας παρουσιάσω τις απόψεις τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράση για το σχέδιο αυτό έκθεση. Συμφωνούμε με πολλά από τα συμπεράσματα της έκθεσης και με την γενική της αξιολόγηση. Σε ό,τι αφορά την εμπορική αυτή συμφωνία θα ήθελα να πω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στις σχέσεις μας με τις δύο αυτές χώρες, Κολομβία και Περού. Το ίδιο θα ισχύσει και για τον, για τον Ισημερινό, το Εκουαδόρ. Ακούστηκαν κάποια πράγματα σήμερα, όπως μια από τις αδυναμίες, αν μπορεί κανείς να τη χαρακτηρίσει έτσι, των εμπορικών σχέσεων μεταξύ Κολομβίας, Περού και του υπόλοιπου κόσμου, που είναι ο μεγάλος βαθμός εξάρτησης από τις εξαγωγές ε, ορυκτών και μεταλλευμάτων. Με τη συμφωνία αυτή θέλουμε να μειώσουμε την εξάρτηση σε λίγες εξαγωγές μεταλλευμάτων. Για την ε, Κολομβία και το Περού τα δείγματα είναι ενθαρρυντικά. Υπάρχουν πολλές έψιλων στις δύο χώρες που αρχίζουν να εξάγουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίω ε, μη παραδοσιακά γεωργικά προϊόντα. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Πρέπει να το τονίσουμε, διότι δεν ξέρω, μπορεί να γιατί μιλάω για κάτι που είναι πιο πολύ στην αρμοδιότητα της ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Trade, εμπόριο. Το λέω γιατί όλα αυτά θα βοηθήσουν την ανάπτυξη περιφερειών, ε, περιοχών στην Κολομβία το οποίο μέχρι στιγμής δεν είχαν τόση πρόσβαση στις διεθνείς αγορές και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, ιδίω ε, στο πλαίσιο της υλοποίηση της Ερνητικής Συμφωνίας ε, της Κολομβίας. Τώρα, δεύτερον, πολλά υπόθηκαν από τους βουλευτές σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα εργασιακά δικαιώματα. Ανησυχίες εκφράστηκαν. Αναφέρθηκε επίσης ο, ακόμη πολύ μεγάλος αριθμός δολοφονιών ε, συνδικαλιστών. Πρόκειται για κάτι που ανησυχεί ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα θέμα που συζητείται πολύ συχνά μεταξύ των Κολομβιανών αρχών ιδίω και των ε, ξεματούχων της Ένωσης εκεί και σε ό,τι αφορά τις πληροφορίες που λαμβάνουμε για την πολιτική του νέου Προέδρου της χώρας ε, είναι ενθαρρυντικά τα μηνύματα. Φαίνεται να το έχει θέσει προτεραιότητα ο Πρόεδρος της Κολομβίας ε, και θα δημιουργήσει, θα χαράξει νέα πολιτική για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Θα παρακολουθούμε την κατάσταση, θα δούμε σε τι θα συνιστάται αυτή η νέα πολιτική. Επίσης, έχουμε τον ε, επίσημο διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τις δύο χώρες, όπου του τίθενται και αυτά τα θέματα. Έχουμε και πιο άτυπες συνομιλίες, όπου επίσης θέτουμε αυτά τα ζητήματα. Και νομίζω ότι με αφότερες τις χώρες έχουμε τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουμε προγράμματα που θα βοηθήσουν να, να ληφθεί υπόψη και να βελτιωθεί η διάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. τα κεντρικά στην έκθεση ήταν η βελτίωση των εργασιακών δικαιωμάτων κτλ αυτά τα θέματα θα μπορούσαν να είναι αντικείμενο προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να υπάρξει ανταλλαγή εμπειριών, ε, βοήθεια, για να μπορούν οι χώρες να εφαρμόζουν καλύτερες πολιτικές. Εμείς στην ΕΕΔ, αλλά και οι συνάδελφοι μας στην Κομισιόν, είμαστε πρόθυμοι να εξετάσουμε τίματα σχετικά, εφόσον αυτά προκύψουν. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον Υφυπουργό Εμπορίου του Περού για τρία λεπτά. Σας ευχαριστώ και καλημέρα σε όλους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω. Σας, σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μας δίνετε να συμμετάσχουμε στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μας δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για κάποιες από τις εξελίξεις ε, όσον αφορά την εφαρμογή της Συμφωνίας Ελευθέρων Εμπορίου μεταξύ Κολομβίας και Περού αφενός και της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης αφετέρου. Αυτή η συμφωνία έχει τεράστια σημασία για την οικονομική μας ανάπτυξη. Μα έχει επιτρέψει να συνεχίσουμε να έχουμε μια διαρκή οικονομική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Γενικότερα ε, να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, να βελτιώσουμε ε, το βιωτικό επίπεδο του πληθυσμού και να μειώσουμε τη φτώχεια. Αυτό το άνοιγμα στις διεθνείς αγορές έχει συνεισφέρει σε σημαντικό βαθμό από το, 2000, ε, το, το 2017 καταφέραμε να μειώσουμε εκείνους που βρίσκονται κάτω από το όριο της φράσης, ε, ε φτώχεια, συγγνώμη, από 49% ε, σε 21% από το, τα τελευταία χρόνια. η συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ένα σημαντικό στοιχείο που συνεισέφερε σε αυτό. Είναι σημαντική γιατί η διμερής σχέση που έχει το Περού με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επιτυχημένη και σημαντική. Ε, το διμερές εμπόριο έχει... Ε, δεν, ήταν, δεν αναπτύχθηκε και τόσο πολύ εξαιτία τη διεθνούς συγκυρία. Ωστόσο, το 2017, ήδη από το 2017, 2007 έχει αυξηθεί. Είχαμε 14% το 2007 και, το 2000, ε, και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο ποσοστό του 11% είναι, έχει παραμείνει λοιπόν σταθερό. Η έκθεση, το προσχέδιο έκθεσης που σας παρουσιάζεται, είναι ένα σχέδιο με το οποίο συμφωνούμε. Θα σταθώ ιδιαίτερα στο σημείο 8 και 9 που αναφέρεται στον εξυγχρονισμό. Ε, στο, όσον αφορά το Περού, τα τελευταία πέντε χρόνια που εφαρμόστηκε πολιτικά η συμφωνία, έχουν προσθεθεί πάνω από 800 νέα προϊόντα τα οποία το Περού εξάγει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και το 98% αυτών των προϊόντων προέρχονται από μη παραδοσιακού τομεί της οικονομίας, δηλαδή εκείνου που έχουν αυξημένη προστιθέμενη αξία. Και το 90% αυτών των εξαγωγών, των νέων εξαγωγών, προέρχονται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μικροεπιχειρήσεις που ξεκινούν να κάνουν και αυτά τις εξαγωγές τους. Είναι ένα τρόπος δημοκρατικοποίησης της ε, περουβιανής οικονομίας, αν θέλετε. Τώρα, όσον αφορά την Κολομβία, αναφέρεται στο σημείο 18 το ζήτημα των επιθεωρήσεων. Μπορώ να σα μιλήσω από την πλευρά του Περού ότι έχουμε κάνει και εμεί σημαντικέ προσπάθειε για να βελτιωθούν οι επιθεωρήσει των χώρων εργασία. Θα ήθελα να σα δώσω ορισμένα στοιχεία. Έχει αυξηθεί ο αριθμό των επιθεωρητών εργασία. Αυτή τη στιγμή έχουμε 300, 360 τέτοιου επιθεωρητέ το 2016 και αυξήθηκε αυτός ο αριθμός έως το 2018. Έχουμε και ένα σχέδιο αύξησή τους ε, που θα τριπλασιαστούν έως το 2020. Το γεγονό ότι θα έχουμε περισσότερους επιθεωρητές στη διάθεσή μας θα βελτιώσει την παρακολούθηση αυτών των απαιτήσεων. Υπάρχει ξεκάθαρη πολιτική βούληση από την ηγεσία του Περού και προσπαθούμε να αυξήσουμε και τον προϋπολογισμό που είναι διαθέσιμος ε, για τις φορολογικές αρχές και προσπαθούμε να καλύψουμε με φορολογικές αρχές όλη, το, όλη την επικράτεια. Καταφέραμε να επίσης ε, και στον ε, τομέα των θεσμικό και στον τομέα των προτύπων για το περιβάλλον να έχουμε σημαντική πρόοδο. Επικυρώσαμε οκτώ από τις συμφωνίες με το Διεθνή Οργανισμό Εργασίας και επίσης ένα σχέδιο δράσης 2018-2021 με τον Οργανισμό Εργασίας. Προσπαθούμε επίσης να εμπλέκουμε ουσιαστικά το, την κοινωνία των πολιτών. Απευθυνθήκαμε στο Συμβούλιο που εκπροσωπεί τους εργαζομένους ήδη από τον Ιούλιο του προηγούμενου έτους και ξεκινήσαμε συνεργασία η οποία ε, διαρκεί ήδη από τότε, προσπαθώντας να καλύψουμε εκείνες τις πρόνοιες της συμφωνίας που αναφέρονται στην συμμετοχή της ε, κοινωνίας των πολιτών, της ε, DAG. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γενικής Διεύθυνσης Trade για τη συνεργασία. Προετοιμάζουμε επίσης και μία αναλυτική έκθεση η οποία θα αναφέρεται στην θέση του Περού όσον αφορά στη συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και πιστεύω ότι με αυτήν θα σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες και θα φανεί πόσο σημαντική πρόοδο σημειώθηκε στο θέμα έτσι ώστε να εκπληρώσουμε και αυτές τις δεσμεύσεις μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον πρέσβη της Κολομβίας για τρία λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ που μας προσκαλέσατε και θα προσπαθήσω να σας παρουσιάσω συνθετικά. Ε, την έκθεση την έχουμε μελετήσει, πήραμε σημειώσεις ε, και επειδή δεν μπορώ να τα καλύψω όλα θα αναφερθώ μόνο γρήγορα γρήγορα σε δύο-τρία σημεία μετά από όσα ακούσαμε. Πρώτα απ' όλα σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της ειρηνευτικής ε, διαδικασίας ε, η νέα κυβέρνηση της Κολομβίας είναι προσιλωμένη στο στόχο της εφαρμογής όπως μας έχει ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν από δύο εβδομάδες συναντηθήκαμε εδώ ο Υπουργός Εξωτερικών, μίλησα με την κυρία Μογκερίνη σε σχέση με την εφαρμογή από τη νέα ε, κυβέρνηση και θα έρθει σε δύο εβδομάδες στι Βρυξέλλε και ο πρόεδρο Δούκε και θα επαναλάβει αυτές τις δεσμεύσει. Φυσικά υπάρχουν κάποιες αποχρώσεις ε, και κάποιε διαφοροποιήσει ό,τι αφορά αυτή τη συμφωνία και θα σας διαθέσουμε πληροφορίες σε εύθετο χρόνο. Ένα συγκεκριμένο ζήτημα το οποίο αναφέρθηκε στι διάφορε παρατηρήσει ήταν εισαγωγέ ε, ή εξαγωγέ, μάλλον πνευματοδών. Ε, και πραγματικά θέλουμε να βελτιώσουμε ε, την κατάσταση. Ό,τι απορία έχετε μπορούμε να τα συζητήσουμε. Πιστεύω ότι οι εμπορικές, ε, πολιτικές, οικονομικές σχέσεις έχουν βελτιωθεί. Είστε ο δεύτερος εταίρος τη εξαγωγής, 14% του συνόλου το 2017 και 15% τρίτη πηγή ε, εισαγωγών. Σε ό,τι αφορά τις ξένες επενδύσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυξήσει τις ε, επενδύσεις το 2017 κατά 40%. Επίσης, έχουμε περιλάβει μη ενεργειακά προϊόντα όπως κακά, τροπικά φρούτα και το αβοκάντο στις εξαγωγές μας και άλλα βιομηχανικά και γεωργοδιατροφικά. Το 78% των εξαγωγών φρούτων από την Κολομβία έχουν προορισμό την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεταξύ των βασικών δικαιούχων και ωφελούμενων από συμφωνία είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, και οι αγρότες μας από 385 δήμους, 32 νομούς, 20 από αυτούς είναι από τις πιο πληγέσες περιοχές από αυτή τη σύγκρουση. Θέλουμε λοιπόν ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει αυτή τη δικασία ε, για την παγίωση της γεωργικής δραστηριότητας και με προορισμό της, πιο πολύ με στόχο της εξαγωγής. Επίσης, νομίζω ότι πρέπει να τονίσουμε σε ό,τι αφορά, ότι ό,τι αφορά τις πολιτικές και τις φυτογενομικές, ε, τους φυτογενομικούς κανόνες, ε, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ε, η επιστημονική γνώση καθώς και το διεθνές δίκαιο. Είναι σημαντικό να έχουμε τεχνική βοήθεια για προϊόντα που προορίζονται για την Ευρωπαϊκή Αγορά, όπω το κακάο, για μα είναι προτεραιότητα για να βγούμε από την κατάσταση καλλιεργειών και εναλλακτική καλλιέργεια. Επίσης θεωρούμε ότι πρέπει να προστατευτούν τα δάση και το περιβάλλον και έχουμε στρατηγική για τον έλεγχο της ε, αποψήλωσης των δασών, για τη διαχείριση προστασία των ευάλωτων περιβαλλοντικών ε, ε, ζωνών. Πρωτοβουλίε για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Επίση, ε, τα γεωργικά όρια τα έχουμε καθορίσει και θέλουμε ε, να προστατεύσουμε επίση προ τα προϊόντα όπω είναι το φινικέλο, ο καφέ, το κακάο κτλ. Τέλο, πρέπει να τονίσουμε τη σημασία του ένα του τίτλου τη συμφωνία που μόλις ε, εκπληρώσαμε. Δηλαδή λειτουργεί πλήρως πλέον ο Εθνικός Μηχανισμός ε, Διαβούλευσης. Έχουμε αναγνωρίσει και ε, την ανάγκη να δημιουργηθεί αυτή η εσωτερική συμβουλευτική ομάδα. Τέλος, θα πρέπει να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε πλήρως όλα τα βήματα της συμφωνίας. Άρα πρέπει να επικυρωθεί πλήρως συμφωνία από τα δύο κράτη που δεν το έχουν κάνει ακόμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Πρέπει επίσης να υπάρξει εξέλιξη στον τομέα της συνεργασίας. Ε, ήταν επομένω θετικά τα πρώτα πέντε χρόνια από την θέση ισχύ τη ε, πολυμερού εμπορική συμφωνία, αλλά χρειάζεται πολλή δουλειά ώστε να έχουμε ακόμα μεγαλύτερη βελτίωση την επόμενη πενταετία. Ευχαριστώ πολύ και τώρα το λόγο κύριο Φίσα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους Σκιώδης αλλά και όλους τους συναδέλφους, καθώς επίσης και τους εκπροσώπους της Κολομβίας και του Περού, να τους ευχαριστήσω για την ε, γενικά θετική υποδοχή αυτής της ε, έκθεσης. Ε, βεβαίως μπορούν να βελτιωθούν περαιτέρω ε, τα πράγματα μέσω τροπολογιών ενδεχομένως. Νομίζω ότι θα πρέπει λίγο να αξιολογήσουμε πού βρισκόμαστε πριν σε σχέση με τις δύο αυτές χώρες και πού βρισκόμαστε τώρα, ε, ποιες είναι οι βελτιώσεις. Ε, νομίζω ότι έγινε μεγάλη πρόοδος λόγω ακριβώς της συμφωνίας, πρόοδος σε οικονομικά αλλά και κοινωνικά ζητήματα νομίζω ότι χωρίς ε, την ε, συμφωνία η κατάσταση θα ήταν πολύ δυνότερη. Οπωσδήποτε θα πρέπει να επαγρυπνούμε, θα πρέπει να συνεχίσουμε την εργατή δουλειά ε, για τα κοινωνικά ζητήματα που είναι φυσικά πολύ σημαντικά και θα ήθελα ε, ε, βάσει και της, ε, πρόταση της πρότασης της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης να υπάρξει μια αρρωγή για ανθρωπιστικά ζητήματα. Να το ξαναδούμε αυτό γιατί οτιδήποτε γίνει κατά την έννοια αυτή μπορεί οπωσδήποτε να είναι ιδιαίτερος χρήσιμο. Να ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά όλους. Περιμένω τα γραπτά σας σχόλια, τις τροπολογίες σας. Ε, έτσι ώστε να έχουμε συνολικά μια καλή ισορροπημένη γνωμοδότηση η οποία θα αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα, τα όσα έχουν συμβεί μέχρι τώρα, αλλά και τις προσδοκίες που μπορούν να έχουν οι χώρες αυτές σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι τις 15 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα θα πρέπει να έχετε υποβάλει τις τροπολογίες σας. Και με τον τρόπο αυτό ολοκληρώνεται η μελέτη του, ε, σημείου 6. Ε, θα διακόψουμε ε, για ένα λεπτό, μια και το σημείο 7 είναι και κλεισμένον των θυρών και επομένως θα πρέπει να εγκαταλείψουν ησύχως την αίθουσα όσοι δεν έχουν δικαίωμα να μείνουν. Και αυτό να το κάνουν όσο γίνεται πιο γρήγορα.